συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο δεν έχετε άλλε παρατηρήσει. Τα ψηφίσματα που υιοθετήσαμε στη σημερινή συνεδρίαση θα προωθηθούν στα αρμόδια σώματα που αναφέρονται στα ίδια τα ψηφίσματα. Διακόπτεται εδώ η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Σα εύχομαι σε όλου καλή επάνωδο.